συνάδελφος Χριστιάνα Μουσκαρτίνη μου διαβίβασε ότι στις 15 Οκτωβρίου προσχώρησε στην ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Ερχόμαστε τώρα στη διάταξη των εργασιών.